Επόμενο σημείο. Δεύτερη ανάγνωση. Τη κοινή θέση όσον αφορά τι καθολικέ υπηρεσίε δικαιώματα των Χριστών Χάρμπορ. Κοινή θέση. Ψηφίζουμε. Κύριε Μάν. Yeah. Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι για την ησυχία στην αίθουσα. Προηγουμένως που έγινε ένα μικρό διάλειμμα κατάφερε κάποιοι κατάφερε κάποια υποψήφια να δημιουργήσει πρόβλημα εδώ στο κοινοβουλίο γιατί μπήκε χωρίς να έχει δικαίωμα να μπει εδώ. Θα το ερευνήσουμε λέει η Πρόεδρος. Thank you very uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ψηφοφορία που θα γίνει. Φαίνεται ότι ψηφίζαμε για το κείμενο της Επιτροπής πριν ψηφίσουμε για τις τροπολογίες. Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο έπρεπε να γίνει, να ξεκινήσουμε από τις τροπολογίες και να ξεκινήσουμε μάλιστα με αυτήν που είναι ε, ε πιο απομακρυσμένη από τη θέση του εισηγητή κτλ. Κυρία Πρόεδρε, χρησιμοποιήστε το άρθρο 19 του κανονισμού και παρακαλώ αν είναι δυνατόν να το προσέξετε ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για δικαιώματα των πολιτών εδώ και για την έκθεση Χάρμπορ και για την έκθεση Τράουτμαν. Πρόεδρος, συγγνώμη, τουλάχιστον για την έκθεση Χάρμπορ ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στο κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν. Πρώτη δέσμη του πακέτου των συμβασμών και το αντίστοιχο κομμάτι που θα ψηφίσουμε στο ένα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αν γίνει ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Όντω εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στο άρθρο 20 με 4 τροπολογίες και το αντίστοιχο τμήμα του 103 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. The others have fallen. Um, we now go to uh, the corresponding part of Amendment 103 by roll call vote. The vote is now open. Ονομαστική ψηφοφορία για το 103 για το αντίστοιχο κομμάτι στο πακέτο. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκατόν ένα. 111, 117. Είναι ταυτόσιμες με νομιστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Και τώρα. 102, 112, 118. Και αυτές με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 62, 94, 104 και 119 που είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Το 96, 106, 120 Ταυτόσιμες. με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Το αντίστοιχο τμήμα το 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η παράγραφος ε, 83, το αντίστοιχο τμήμα του 103, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, η τελογική 26 και το αντίστοιχο τμήμα του 103, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 18. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. απορρίπτονται 95, 105 και 114. Είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Εγκρίνεται από σε κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε. επόμενο ε, θέμα είναι σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έκθεση Τράουτμαν ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ζήτησα το λόγο επειδή δεν συμφωνώ με τη σειρά γιατί στην ψηφοφορία της έκθεσης Τράουτμαν. Πριν από τη συμβαστική λύση 10 θα ήθελα για να εξηγήσω περαιτέρω να μου δώσετε το λόγο. Πριν να ψηφίσουμε τη συμβαστική λύση 10. Πρόεδρος, ναι, ωραία, για την... Ε, ε θα σας ακούσουμε τότε όταν φτάσουμε στη 10. Ωραία. Μπλοκ παριθμών 1, συμβεβασ... ε, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνονται. Τροπολογία, τροπολογίες 3 και 7, ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτονται. Το αντίστοιχο σημείο της τροπολογίας ένα, λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Okay. Mrs. Harms. Κυρία Harms. θα ήθελα να ζητήσω εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας να αλλάξουμε τη σειρά της ψηφοφορίας. Υπάρχουν ψηφοφορίες που μοιάζουν μεταξύ τους από διάφορες πολιτικές ομάδες. Αυτές θα πρέπει να τις ψηφίσουμε πριν φτάσουμε συμβαστική ψηφο... στην τροπολογία 10. Γιατί το λέω αυτό, γιατί... Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών για την πρόσβαση στο διαδίκαιο, αυτά είναι αυτό είναι ένα θέμα που ξεπερνάει πολύ περισσότερο την τροπολογία και βεβαίως θα θυμάστε την τροπολογία Μπόνο Bendit εκείνη η τροπολογία έκανε θόρυβο, πάταγο και θα πρέπει να τονίσουμε και τούτην εδώ την πρωτολογία, τροπολογία η οποία αναφέρεται και πάλι στο ίδιο θέμα, στα δικαιώματα του πολίτη σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η... Νομίζω ότι τα καλά αποτελέσματα της δέσμης Telecom δεν ε, είναι ότι δεν πρέπει να το χαιρετήσουμε αλλά δεν θα πρέπει τελικά να μας οδηγήσει στο να αγνοήσουμε δικαιώματα πολιτών σαν και αυτά που περιέγραψα εγώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, βάσει του 154 και συγκεκριμένα της παραγράφου 2 συμφωνούμε με και αυτό που ζητήθηκε να αλλάξουμε τη σειρά των ψηφοφοριών να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες 1, 2, 5, 6 και 9 πριν από την τροπολογία τη συμβεβαστική 10 χτες η Βεβαίω πάρθηκε η απόφαση στην πολιτική μας ομάδα ότι θα υποστηρίξουμε τη συμβιβαστική λύση 10 αλλά ε, εν πάση περιπτώσει εμείς ζητούμε να αλλάξει σειρά των ε, ψηφοφοριών και ε, δεν θα υπερψηφίσουμε τη συμβαστική λύση 10 γιατί θα, κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση πριν να επιμείνουμε για αλλαγή της συμπεριφορά των πολιτών κτλ. Ε, κυρία Πρόεδρε ζήτησε το λόγο όχι ε, σαν πρόεδρος της ε, οποιαδήποτε επιτροπής αλλά σαν ε, εισηγήτρια για την ομάδα μου για το θέμα για την έκθεση Τράουτμαν αγαπητοί συνάδελφοι κανείς εδώ σε αυτό το όργανο δεν θέλει να περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το έχουμε πει επανειλημμένο, το έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένο με τη Τσεχική Προεδρία. Όλε οι πολιτικέ ομάδε, όλα τα πολιτικά κόμματα συμμετείχαν στις συζητήσεις αυτές. κανεί, δεν θέλει να περιορίσει τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με το διαδίκτυο. Γι' αυτό σα παρακαλώ να μην συμφωνήσετε με την ανατροπή τη σειρά των ψηφοφοριών, να διατηρηθεί η σειρά των ψηφοφοριών ψηφοφοριών ως έχει. Πρόεδρος, η κυρία Τράουτμαν ως εισηγήτρια θέλει το λόγο. Ναι κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να πω σχετικά με το αίτημα αλλαγή ε, της σειράς ε, στο κατάλογο των ψηφοφοριών. Αν ο... <laughs> Αν ο συμβιβαστική αυτή λύση μπήκε πριν από τις τροπολογίες των ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων αυτό συνέβη επειδή βρίσκεται πιο μακριά από τη δική μου την έκθεση από ότι οι τροπολογίες των πολιτικών ομάδων περιλαμβάνει πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούν έως και να επηρεάσουν κάποια δικαιώματα χρηστών. Επίσης, για το άρθρο 1 που αφορά στο πεδίο εφαρμογής ε, ε, αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η τροπολογία 10 ενώ οι τροπολογίες των πολιτικών ομάδων είναι πιο συγκεκριμένες και αναφέρονται στους εθνικούς, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Θα ήθελα επίσης να πω κυρία Πρόεδρε ότι έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις. Ξέρω ότι μια ομάδα ε, αυτή τη στιγμή... άκουσα ότι μια ομάδα δεν θα υποστηρίξει πλέον τη συμβαστική αυτή τροπολογία και γι' αυτό και έχω πάρει θέση για τη συμβαστική αυτή λύση όπως έχω πάρει θέση και για την ανθρωπολογία 46 υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες συζητείτε το θέμα αυτό καλύτερα η Ολομέλεια να ακολουθήσει την δεδομένη σειρά που υπάρχει εδώ και να μην πάρει ε, θέση για ένα θέμα το οποίο ενδεχομένω θα επανέλθει στο, στην Ολομέλεια. Ε, αν ε, Λοιπόν, εάν ε, επίση συμβούν ορισμένα πράγματα, αν υπάρξει ανατροπή, αν θέλετε, τη ψηφοφορία ή ε, το αποτέλεσμα τη 46 είναι quarante six n'obtient pas la είναι υπέρ τότε δεν αλλάζει τίποτε αν όμως η, καταψηφιστεί η 46 τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική λύση την ε, τροπολογία 10 δηλαδή πρόεδρος άκουσα τις απόψεις διαφόρων και έλαβα υπόψη μου και αυτό που είπε η συγγήτρια. Συμβουλεύτηκα και τις αρμόδιες υπηρεσίες και άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά που ελέγχθη. Ως πρόεδρος βάσει του 155.2 του κανονισμού έχω το δικαίωμα να αποφασίσω τη σειρά των ψηφοφοριών. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό και στο ιστορικό αλλά και στο εξωτερικό αυτού του οργάνου ε, ε, που θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, και ε, να ψηφίσουμε πρώτα για τις προηγούμενες τροπολογίες. Εξ όσων γνωρίζω, η τροπολογία 10 κατετέθη μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω γιατί πρέπει να ανατρέψουμε τη σειρά των ψηφοφοριών, να αλλάξουμε τη σειρά των ψηφοφοριών. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινώ. με τις τροπολογίες 1, 2, 5, 6, 9 τα αντίστοιχα μέρη τους ε, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Is ψηφίσατε όλοι The vote is now closed. Πέρας της ψηφοφορίας It is adopted και εγκρίνεται, εγκρίνονται. Amendment 4, I put amendments... Τροπολογίες 4 και 8 με ονομαστική ψηφοφορία. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτονται. Η κοινή θέση λοιπόν εγκρίνεται έτσι όπως τροποποιήθηκε. Το επόμενο θέμα είναι σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση φορέας προβαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσία. Ψηφίζουμε σχετικά με την κοινή θέση Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η κοινή θέση λοιπόν εγκρίνεται ως τροποποιήθηκε. Mrs. Troutman κυρία Τρότμαν. Κύριε Πρόεδρε, Είχα ζητήσει να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και για την συμβιβαστική, γιατί ήταν μια συμβιβαστική που ήταν, ε, είχε μεγαλύτερο, ευρύτερο μάλλον πεδίο από ότι η τροπολογία 46. Δεν, δώσατε, δεν βάλατε στην ψηφοφορία τη συμβιβαστική χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση, ούτε ε, ε, σχόλιο στον εισηγητή και λυπούμε που δεν ακολουθήσατε την ε, σύσταση της ε, εισηγήτρια για την ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια. Να πω επίσης και να εξηγήσω την ψηφοφορία που μόλι έγινε ότι από τη στιγμή που οποιοδήποτε μέρος του συνόλου της συμβιβαστική δεν έχει οθετηθεί, το σύνολο του πακέτου θα πάει στη συνδιαλέγη. Αυτή είναι η συνέπεια των όσων έγιναν σήμερα. Σας ευχαριστώ κυρία Τρότμαν. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουν τις συνέπειες των όσων ψηφίζουν. Έχετε δίκιο, αλλά δεν, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε στην άλλη συμβιβαστική και ούτως ή άλλως η ψηφοφορία ήταν σαφέστατη. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για την έκθεση ε, Γκουεζέλο Ζαγκηγιάρ για τη ζώνη συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές ε, τηλεπικοινωνίες ε, με επίγεια βάση. Τροπολογία 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε τώρα. Everybody Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας ε, Λούλη για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Τροπολογίες από την αρμόδια επιτροπή είναι 21 τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, Θα ήθελα να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ για την τροπολογία 20 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Τροπολογίες 21. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να το ελέγξουμε, γιατί δεν σηκώνετε όλα τα χέρια σας. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την 21, τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 26, 36, ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, να το ελέγξουμε. 36 λοιπόν ψηφίζουμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 13 και 39 μαζί. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω πως η κυρία Λούλινγκ θέλει να κάνει μια προφορική τροπολογία. Κυρία Πρόεδρε, έχω συμφωνήσει με τον κύριο Κοτσλόβο που ήταν ο εισηγητής για τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Απασχόληση ώστε να εντάξουμε σε αυτό το σημαντικό άρθρο 6 την εξή ρήτρα. Αν η νομοθεσία ενός κράτους μέρους δεν προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη του ανεξάρτητου επαγγελματία στο καθεστώ κοινωνική ασφάλιση, αυτή δίνεται υπό κατόπιν αιτήματο ε, του συζύγου βοηθού. Θέλουμε δηλαδή υποχρεωτικά να ασφαλίζεται και ο σύζυγο, όπω συμβαίνει και για του ανεξάρτητου επαγγελματίε. Αν όμω σε κάποια χώρα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για του ανεξάρτητου επαγγελματίε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε να γίνεται αυτό υποχρεωτικά για του συζύγου. Και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε αυτή την παραπάνω, το παραπάνω εδάφιο. Και υποβάλλω αυτή την προφορική τροπολογία και εξ ονόματος του κύριου Κοτσιλόβου. Υπάρχουν εδώ αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις. 40 πρέπει να είναι αντίθετη. Έχουμε 40 που είναι αντίθετοι, οπότε φοβούμαι, κυρία Λόλινγκ, που δεν θα υποβληθεί αυτή η τροπολογία. Δεν θα ψηφιστεί η προφορική σα τροπολογία. Θα ψηφίσουμε σε τέσσερα τμήματα την τροπολογία 14. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξω, αν θέλετε. Αρχίζουμε έλεγχο λοιπόν για τη 42. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για δύο ψήφους. 16. Ψηφίζουμε την 16. Υπέρ, κατά. Αποχές. We will check it. Amendment 16, if we open the vote, please. Το ελέγχουμε. Τροπολογία 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Everybody voted. The vote is now closed. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Λούλινγκ. Προχωράμε στη ψηφοφορία για την έκθεση Εστρέλα. για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας και την εργασία των εγγύων, λεχώνων και γαλαχουσών εργαζομένων. Η κυρία Στρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τις υπηρεσίες να προσέξουν ότι η γλωσσική εκδοχή που ισχύει για όλες τις τροπολογίες είναι η πορτογαλική. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να ζητήσω η σειρά της, τροπο, ψηφοφορίας να αλλάξει η τροπολογία 43 της Επιτροπής να ψηφιστεί πριν από την 83 για λόγους ε, συνέπειας συνοχής. Τέλος, να θυμίσω ότι η οδηγία αυτή που θα τροποποιήσουμε είναι ήδη 17 χρονών είναι ήδη δηλαδή υπεπαλαιωμένη, ε, απαρχαιωμένη. Η αναθεωρημένη οδηγία δεν θα αρχίσει να ισχύει παρά μετά το τέλος της επόμενης θητείας. Δηλαδή νομοθετούμε για το μέλλον, όχι για το παρόν. Και κυρίως νομοθετούμε για το καλό των, πολίτων, ε, των πολιτών, γιατί υπάρχουν, ε, μάλλον έτσι τους δίνουμε περισσότερους λόγους για να ψηφίσουν τον επόμενο Ιούνιο. Να ολοκληρώσω ζητώντας τη στήριξη των συναδέλφων για την ε, έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Λούλινγκ. Κυρία Πρόεδρε, επειδή τα πράγματα είναι όπως είναι για αυτήν εδώ την έκθεση. Υπάρχουν 89 τροπολογίες. Είναι πραγματικά χαοτική η κατάσταση και η ψηφοφορία που θα κάνουμε δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε πραγματικά μια αντικειμενική συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Υπάρχουν 89 τροπολογίες οι οποίες είναι τελείως αντιφετικές οι δε. Γι' αυτό προτείνω εγώ την ε, παραπομπή αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή γιατί όπως είπε και η κυρία Εστρέλα έχουμε και χρόνο. Πολύ. Κυρία Λούλινγκ, αυτό το αίτημα το κάνατε εξ ονόματος πολιτικής σας ομάδας. Μάλιστα, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Όχι. Δεν κάνω ποτέ τίποτα που να μην είναι εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας. Όχι, απλώ ήθελα να το καταλάβω για να δω τι θα κάνω με το έτοιμά σα. Επειδή κάνατε εσεί ε, το έτοιμα της παραπομπής, θα εξετάσουμε αυτό κατά προτεραιότητα. Υπάρχει κάποιο άλλο υπέρ αυτή τη πρόταση. Όχι. Κατά? Όχι. Ωραία. Να το ψηφίσουμε τότε. Ποιοι είναι υπέρ μιας παραπομπής στην Επιτροπή. Κυρία Στρέλα, φαίνεται να ζήτησε το λόγο και ως εισηγήτρια νομίζω θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να μιλήσει. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχει νόημα να παραπέμψουμε στην Επιτροπή και πάλι αυτή την έκθεση, γιατί συζητήθηκε με όλες τις ομάδες Υπάρχει η στήριξη που εγώ θεωρώ πώ είναι πλειοψηφία σε αυτή την αίθουσα. Συζητήθηκε με, στην με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές θέσει. Εμείς γνωρίζουμε ότι δυστυχώς το Συμβούλιο υπό την Τσεχική Προεδρία ε, είχε μία πολύ συντηρητική στάση γιατί δεν θέλησε να προωθήσει την ισότητα των φίλων και πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να υποστηρίξουμε αυτές τις προτάσεις να είναι καλύτερη η έκθεση γιατί έτσι όπως σας είπα θα έχουν περισσότερους λόγους οι πολίτες μας να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Σας ευχαριστώ κυρία Εστρέλα. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την πρόταση της κυρίας Λούλινγκ και του ΕΛΚ για παραπομπή στην Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγώ νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά ευχαρίστως να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την πρόταση της κυρίας Λούλινγκ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας και σαφώς εγκρίνεται η παραπομπή στην Επιτροπή. Η Έκθεση επόμενη είναι η έκθεση της κυρίας Στάουνερ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση Επιτροπής ε, όπως προποποιήθηκε, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στην εισηγήτρια. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Μαλντίκη για το πρόγραμμα στήριξη οικονομική ανάκαμψη μέσω χορήγηση κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση σε προγράμματα στον τομέα τη ενέργεια. Ψηφίζουμε το, το πρώτο σύνολο τροπολογιών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, το δεύτερο πακέτο ε, καταπίπτει, τροπολογία 13, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τρο... πρόταση όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική και ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. κύριος ε, Μπέγκη νομίζω έχει μια προφορική όσον αφορά το σχέδιο ψηφίσματος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σε συνεννόηση με τον εισηγητή Μαλνταϊκές οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του νομοθετικού ψηφίσματος τροποποιήθηκαν και για το παράγραφο 2 πρέπει να πούμε ότι το ποσό το αναφοράς η, πρέπει να αντιστοιχεί όπως αναθεωρήθηκε και μετά στο 3 διαγράφεται η πρώτη πρόταση και στην παράγραφο 5 λέμε ότι η νομοθετική διαδικασία εκπληρώθηκε μετά την χρηματοδότηση του προγράμματος. Έχετε ενστάσεις. Όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου που χρησιμοποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση Κάρας για τις ε, τράπεζες και συνδεόμενα ε, ε και συνδεόμενες και, και κεντρικές τράπεζες το... η έκθεση αυτή είναι αρκετά αμφιλεγόμενη και για να είμαστε δικαιοί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας είναι, θα ήθελα να μου δώσετε το λόγο πριν από την αιτιολογική έκθεση 3. Πρώτο μπλοκ. το αντίστοιχο τμήμα είναι υπέρ, είναι κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90, μυρομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. That is rejected. We now therefore go to amendments 88 and 93. 88 και 93 που είναι ταυτόσιμες με Τώρα ψηφίζουμε. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και απορρίπτονται. Και πάμε στο 81 μοιρομαστική. Ψηφίζουμε. Η τροπολογία 91. Ψήφισαν όλοι. Vote is now ε, απορρίπτονται και αυτές και τώρα πάμε στο αντίστοιχο τμήμα της 89. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο κύριος Μπούλμαν ζητεί το λόγο Κυρία Πρόεδρε για το βασικό κεφάλαιο πρόκειται εδώ και οι τροπολογίες 92 και 91 ε, είναι ε, εκείνες οι οποίες μας επιτρέπουν να, έχουμε την σαφέστερη ε, ρύθμιση του θέματος γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να ψηφίσουμε πρώτα 92-91 και μετά την 89 ε, με την μορφή του εκτιμώντα του αιτιολογικής σκέψης 3. Πρόεδρος, για να δούμε με ποια σειρά θα τα κάνουμε. Ε, το διαδικαστικό κύριε Κάρας που είστε ο συγητής. Ναι, θέλω να πάρω το λόγο, λέει ο κύριος Κάρας, γιατί έγινε συζήτηση και διαπιστώσαμε ότι η και ότι οι τροπολογίες ρυθμίζουν ορισμένα πράγματα ε, με αρκετή λεπτομέρεια να παραμείνουμε στη σειρά που έχει οριστεί τώρα και για την ονομαστική ψηφοφορία δεν έχω τίποτα να πω. Έχετε κάποια ένσταση όσον αφορά το αίτημα για ονομαστική. Όχι. Ο, άρα ε, θα κάνουμε αυτό το οποίο με, με αυτή τη σειρά, με το διαδικαστικό. Και έχουμε τώρα τις τροπολογίες. 86 και 87 έχουν όμω ε, αποσυρθεί και τώρα πάμε στο αντίστοιχο τμήμα του 89 την υπέρ ονομαστική, συγγνώμη. Ψηφίζουμε τώρα στον αντίστοιχο τμήμα του 89. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνονται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το υπόθεση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε πει είναι υπέρ είναι κατά αποχές εγκρίνεται και το σύνολο της νομοθετικής πρότασης με ονομαστική ψηφίζουμε τώρα Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, εισηγητά. Το επόμενο θέμα θα ψηφίσουμε την έκθεση Χόπενστεντ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναφορά και έλεγχο. Το πρώτο μπλοκ, πίνει υπέρ, πίνει κατά. Αποχές, εγκρίνεται. πρόταση της Επιτροπής όπως τοποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σχέδιο του ψηφίσματος ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται και συγχαρητήρια σε Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Βοητσιετσόφσκι για την προστασία των ζώων την ώρα της σφαγής. Θέλει τον λόγο ο κύριος εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο σύντομες αλλά σημαντικές τεχνικές ερωτήσεις. Έχουμε ένα μπλοκ τροπολογιών από την Γεωργική Επιτροπή μεταξύ των οποίων και το 64 θα πρέπει να γίνει χωριστή ψηφορία τούτων αφορά το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς που το πρέπει να συγκροτηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό με του κανονισμού. Η Επιτροπή Γεωργίας λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η υποχρέωση του να φτιαχτεί ένα τέτοιο κέντρο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο κατά γνώμη μου όσοι συγκριτούν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει προς το όλο πνεύμα του κανονισμού. Το 64 να ψηφιστεί χωριστά παρακαλώ. Δεύτερο θέμα θέλω να σας αναφέρω, παρακαλώ, προσέξτε το 28. Μιλά για αυτό το φορτισμένο ζήτημα της τελετουργικής θανάτωσης. Εάν ψηφίσουμε υπέρ, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα απαγόρευσης τέτοιας θανάτωσης σε εθνικό επίπεδο. Εάν καταψηφιστεί αυτή η τροπολογία το 28, τότε θα είναι δυνατόν να επιβάλλεται τέτοια απαγόρευση. Επίσης, προσέξτε το 85. Λέει η Κομισιόν ότι θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς των ζώων από την εκμετάλλευση στο σφαγείο και να πάμε στις 24 ώρες. Εάν το 85 εγκριθεί, δεν θα έχουμε τη μείωση του χρόνου μεταφοράς. Εάν καταψηφιστεί η τροπολογία, το 85, θα στηρίξουμε την Κομισιόν όσον αφορά τη μείωση του χρόνου μεταφοράς. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Για το 64 και το 17. Υπάρχει κάποια ένσταση σε αυτό που μας είπατε. Οπότε συνεχίζουμε με την ψηφοφορία όπως προβλεπόταν να γίνει. Και θα ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες αρμόδιας επιτροπής θέση 69 ψηφίζουμε. Εγκρίνονται 69 τροπολογίες. Τροπολογία 2, ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται 15 με ονομαστική ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας 20 με ονομαστική ψηφίζουμε το 20 ψήφισαν όλοι πέρας 21 με ονομαστική. Ψηφίζουμε το 21. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται η 28 με ονομαστική. Ψηφίζουμε το 28. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 37 ή ονομαστική. Ψηφίζουμε. Το 37. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 50. Ψηφίζουμε. Επί του 50. Ψήφισαν όλοι. Τέλος και εγκρίνεται. 51. Ψηφίζουμε με ονομαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική. 52. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 87, ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 93, με ονομαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 ονομαστική ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος αφού θέλετε για το 100. Όλοι ψήφισαν. Πέρας. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 θα πρέπει να γίνει έλεγχος ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Σαράντα επτά, πέρ, κατά. Εποχές, Απορρίπτονται. 121 υπέρ κατά εποχές δεν γίνεται 124 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 103 υπέρ εγκρίνεται το 59 καταπίπτει και πάμε στο 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα του 105 καταπίπτει και πάμε στο αντίστοιχο τμήμα του 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 106 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, θα ελέγξουμε την 85 ηλεκτρονικά. Σφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 125 κατά πίπτη, 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117. 118 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Τροπολογία 4, ονομαστική. Ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, το σύνολο της προτάσεως Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφίστε παρακαλώ ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για την έκθεση Χωσέ Αλμπίνο Σίλβα Πιναϊδα για την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Παράγραφος 14. Δίνω το λόγο στον κύριο Πουσομάσιος. Ναι κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα και θα ε, ήθελα να με συγχωρήσει το σώμα για μια τελευταία προσωπική πα, τροπολογία που θα κάνω. Υπάρχει, πρόκειται για δύσκολο θέμα, οι μετάφραση διάφορες γλώσσες δεν είναι πάντα καλή. Αντί για την παράγραφο 14 έτσι όπως έχει γραφτεί να αυτή να αντικατασταθεί από την παράγραφο 3 της, του ψηφίσματος της 11ης Τρίτου 2009 ε, που σχετιζόταν με το Ιρανικό ε, Αρινό Συμβούλιο για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Λέει κάποια κράτη-μέλη έχουν εισάγει την έννοια του κατώτατου μισθού και ζητεί από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τηρήσουν τις προϋποθέσεις για την σωστή ίση συμμετοχή όλων και να μην και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αν θέλουν του κατώτερου μισθού των κοινωνικών διαπραγματεύσεων συλλογικών διαπραγματεύσεων κτλ. Ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δέχτηκαν όλες οι πολιτικές ομάδες και ο εισηγητής συμφωνεί με αυτό. Ελπίζω λοιπόν το Σώμα να επιτρέψει την ε, κατάθεση αυτής της τρο, προφορικής τροπολογίας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Αντιδράσεις υπάρχουν. Ο κύριος Άντερσον ζήτησε το λόγο. Tack så mycket. Bara en kort upplysning om den svenska översättningen. Nej, Για την paragraf 3 άκουσα να λέγεται ότι το ελάχι, να, κατώτατο μισθό να μιλάτε αλλά πρόκειται για το ελάχιστο εισόδημα άλλο το εισόδημα και άλλο η, η και άλλο κατώτατος μισθός διόρθωση να γίνει για το 13 και το 36 μάλιστα να πω και εγώ ότι δεν υπάρχουν λοιπόν τώρα ε, λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 36 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο με προονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Λαμπέρ για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. I would check it if you Ωραία, να το ελέγξουμε. So if we can Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται Κατά εξαίρεση προς τη συνήθεια δικασία Αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν διευκρινήσεις ε, ψήφου, επειδή ε, έχουμε αργήσει πολύ, το... Υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος αριθμός διευκρινήσεων ψήφου. Δεν θα μπορέσουμε ούτε μέχρι τις 3 να τελειώσουμε. Γι' αυτό παίρνω την απόφαση όπως έχει και στο παρελθόν ε, να γίνουν οι διευκρινήσεις ψήφου στο τέλος των εργασιών απόψε. Tonight. Ωραία, μία διευκρίνηση ψήφου. Τέλο πάντων, φαντάζομαι ότι όλοι θα πείτε το ίδιο. Ναι, οι, οι κανόνε είναι σαφεί. Μετά την ψηφοφορία μπορούμε όλοι να κάνουμε διευκρίνηση ψήφου. Ξέρω ότι έχουμε αργήσει. Γι' αυτό προτείνω μια συμβαστική λύση που είχε χρησιμοποιήσει ο κύριο Κουάδρας όταν έγινε αυτό. Ε, ε, ε, να ακολουθήσουμε τη μέθοδό του για να γίνει αυτή η διευκρίνηση ψήφου ε, προσωπικά η μια μετά την άλλη. Ό, όχι λέει η πρόεδρος, το σκεφτήκαμε αυτό αλλά δεν γίνεται. Ε, το βράδυ, το βράδυ ε, θα δοθούν οι διευκρινήσεις ψήφου.